για την παρουσία σας. Δεν είναι πάντα εύκολο τη Δευτέρα. Είμαστε όμως έτοιμοι για τρεις ώρες συνεδρίαση, έτσι. Ελπίζω να είστε έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι. Να ξεκινήσουμε με την ημέρηση διάταξη, το πρώτο σημείο. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Τώρα, οι ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3, λοιπόν. Ενδιάμεση έκθεση για το πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Θέση του Κοινοβουλίου εν ώψη Θα θέλαμε να συζητήσουμε λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Εγώ είμαι ο εισηγητής στην προκειμένη περίπτωση. Κάποιοι συνάδελφοι και είναι εδώ μαζί μας. Να σας πω ότι έχουμε περίπου μισή ώρα για τη συζήτηση αυτή, λίγο περισσότερο και μάλλον θα χρειαστούν. Συμφωνήσαμε μεταξύ των συντονιστών και σχεδόν εισηγητών σε ό,τι αφορά τη θέση μας ως Επιτροπή Ήτρε, θέλω να υπογραμμίσω τρία γενικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμφωνήσουμε γύρω από μια σαφή μεθοδολογία ε, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία με βάση ε, σταθερές τιμές. Και εδώ συμφωνούμε και με τους συναδέλφους ε, ε, από τη Δημοσιονομική Επιτροπή για να στείλουμε ένα σαφές, καθαρό μήνυμα χωρίς να υπάρχει περιθώριο χειραγώγησης. Και επίση χρειαζόμαστε μια νομικώ δεσμευτική, υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού προγράμματο. προγράμματος, με ρόλο βέβαια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι γενικά ε, σχόλια. Ε, έχουμε την ορίζοντα Ευρώπη. Εμείς είχαμε προτείνει 180 δις. Εξακολουθεί να ισχύει αυτή η πρόταση. EU Invest. έρχονται να προσθεθούν αυτά στο, στο ορίζοντα Ευρώπη. Και αυτό παραμένει η πρότασή μας. Το Connecting Europe Facility. Ε, συνέργειες, όπως αναφέρω την διάμεση ε, έκθεση, είναι υπεραπαραίτητες απαραίτητες συνέργειες αυτές και επιπλέον ε, χρηματοδότηση αποκλειστικά για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης ε, στα πλαίσια του νέου πολιτικού του δημοσιονομικού προγράμματος ε, για τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη χρήση άνθρακα. 13 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία το μεσημέρι για την υποβολή των τροπολογιών. Κάποιες σκέψεις τώρα για τη θέση της Επιτροπής μας, της γενικότερα τη γενική θέση της Επιτροπής μας μάλλον, ε, για τον προπολογισμό στην Επιτροπή Ήτρε θέλουμε να ψηφίσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Ο συντονισμό όμως, επειδή πρέπει να συνεργαστούμε και με την Μεσονομική Επιτροπή και οι συνάδελφοι από την Μεσονομική Επιτροπή, οι συγκητές, οι συντονιστέ, προτείνουν να ορίσουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για τους οικονομικούς φακέλους για τα διάφορα προγράμματα 2021-2027 τεχνική μετάφραση, ουσιαστικά μεταφορά των στοιχείων του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτά τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στο δημοσιονομικό ε, και στην ενδιάμεση έκθεση και στην μελλοντική νομοθετική έκθεση για τα προγράμματα αυτά. Είναι σημαντικό αυτό. Να σας πω τι λένε εδώ οι συνάδελφοι από τη Δημοσιονομική Επιτροπή, τι προτείνουν. Θέλουμε να συμφωνήσουμε πρώτα για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικά και για το σύνολο του οικονομικού φακέλου και στη συνέχεια να δούμε τις ε, νομοθετικές εκθέσεις για τα επιμέρους προγράμματα. Ζήτησα από τους ε, ε, εισηγητές, τους βοηθούς εισηγητές, ε, να αντιδράσουν στη δημοσιονομική πρόταση, να δράσετε λοιπόν ως εισηγητές επί των δημοσιονομικών προτάσεων και με βάση τη, δική σας αντίδραση θα ε, μάλλον μια απάντηση την οποία στείλαμε χθες. Ως ε, ε, εισηγητής της Επιτροπής Ήτρε θα συνεχίσω να συντονίζω τις προσπάθειές μου με τους εισηγητές του, ε, της δημοσιονομικής ομάδας, της ομάδας ε, δημοσιονομικών θεμάτων για την διάμεση έκθεση. Από την Δημοσιονομική Επιτροπή λοιπόν αλλά και με όλους τους κοιόδους συγγητές ε, ε, εγώ θα συντονιστώ. Ήθελα τώρα να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο από τις πολιτικές ομάδες. Ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόταση αυτή της γνωμοδότησης που είναι εξαιρετική βάση συζήτησης τα σημαντικότερα σημεία τα οποία αναφέρατε βεβαίως μας βρίσκουν σύμφωνος. Πρώτα από όλα οι νέες πρωτοβουλίες πρέπει βεβαίως να πλαισιωθούν με νέα και επαρκή κονδύλια. η τα κράτη-μέλη αλλιώς πρέπει να μας πούν από ποιες πρωτοβουλίε, πρωτοβουλίες, ε, πρωτοβουλίες δεν χρειάζονται πια στο μέλλον για να τις ε, περικόψουμε. Ε, γιατί βεβαίω ε, τα προβλήματα αυτά ήταν αυτό το οποίο λέγαμε στα γερμανικά το επισκεπτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλετε το, αυτό το οποίο ακριβώς παρουσιάζει την προσθέμενη αξία της και δείχνει το τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον και νομίζω ότι αυτό πρέπει να παραμείνει έτσι και αυτό εδώ πέρα Συμφωνούμε ακριβώς, ε, κύριε Βούζεκ ότι πρέπει να ζητήσουμε νέα επιπρόσθετα κονδύλια που πρέπει να παρουσιάζονται πάντα σε σταθερές ε, τιμές για να υπάρχει μια συγκρισιμότητα. Γιατί αν ασχοληθεί κανείς να δείτε τι προτείνει η Κομισιόν, ε, βλέπει ότι τα νούμερα είναι ονομαστική αριθμή και όχι αποπληθωρισμένη. Οπότε είναι κάπως ε, αδιαφανή τα νούμερα αυτά. Περισσότερα κονδύλια για τον ορίζοντα Ευρώπη πρέπει να δοθούν, πράγματι. Αυτό σημαίνει ότι εγώ και η ομάδα μου τα 20 δισεκατομμύρια αυτά στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα τα υπερασπιστούμε οπωσδήποτε και γι' αυτό ακριβώς είναι ακριβώς απαραίτητο να δούμε τις ε, παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή. Και είναι σημαντικό για εμάς ακριβώς να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών προγραμμάτων γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένας κίνδυνος μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θεωρώ ότι ο ορίζον πρέπει να παραμείνει πολιτικό έργο και να το πω αλλιώς αν υπάρχει πολιτική βούληση για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, θα πρέπει να ισχύσει πάλι αυτό το οποίο είπα. Επιπρόσθετες αρμοδιότητες πρέπει να σημαίνει επιπρόσθετα κονδυλία και χωριστά από τον ορίζοντα. Οπότε εγώ έλεγα ότι θα προτείνουμε και κάποιες τροπολογίες θα τονίσουν αυτή την ανάγκη ακριβώς για επαρκή κονδυλία στο πει, στα σημεία που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας πρόγραμμα το Διεθνικό ψηφιακή Ευρώπη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγαπητέ συνάδελφοι αν μου επιτρέπετε ε, συντομεύεται δύο-τρεις προτάσεις ακόμα Κύριε Μπούζεκ, καμιά φορά είναι περίπλοκα αυτά τα πράγματα και ίσως να μας δίνετε ένα λεπτό ακόμα. Τέλος πάντων, ολοκληρώνω. Να πω ότι είναι σημαντικό να δοθούν επαρκή κονδύλια για την καταβολήμηση της κλιματικής αλλαγής ε, και υπάρχουν κάποια πολιτικά προβλήματα τα οποία είχαμε δει και στο παρελθόν περισσότερα κονδύλια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεσματική ενέργεια και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ. Και αναμένουμε και τις τροπολογίες σας. Από το ECR, παρακαλώ. εκπροσωπείται από τον κύριο Τσέσακ, ο οποίος αντικαθιστά τον καθηγητή Κρασνοντεύσκη. Δεν μπόρεσε να είναι εδώ και γι' αυτό ο κύριος Τσέσακ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όπως ε, σωστά είπατε, αντικαθιστώ τον καθηγητή Κρασνοντεύσκη και μιλώ εξ ονόματός του καθώς σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, εκ μέρους του κ. Κρασνοντεύσκη για το σχέδιο γνωμοδότησης. Η διατήρηση του προπολογισμού της ΙΤΡΕ είναι πολύ σημαντικό εν ώψη των περικοπών. Η ΙΤΡΕ είναι μια, μια επιτροπή που διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των κοινωνικών αναγκών και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό. Το πρώτο μου σχόλιο έχει να κάνει με το Ταμείο ε, Μετασχηματισμού της Ενέργειας. Ε, και αναφέρομαι σε περιοχές ε, όπου κυριαρχούν οι, τα εργοστάσια ηλεκτρισμού. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη μετάβαση στην αγορά ενέργειας. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπία στην αγορά εργασία. θα πρέπει να προστατεύσουμε τι θέσει εργασία και να δημιουργήσουμε νέε σε αυτέ τι περιοχές. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά το νεοπολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς αυτά τα θέματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη ε, στο μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη θα πρέπει να προβλέπονται και κονδυλία και για την υποδομή αερίου συγκεκριμένα εν ώψη των περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, μεταφορά ε, κονδυλίων μεταξύ των διάφορων ταμείων. Αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ των κρατών μελών και αν και καλωσορίζουμε τον ε, κανονισμό περί κοινών διατάξεων, Πιστεύουμε ότι αυτό το μέσο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν τα εθνικά κονδύλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, μίλησατε τους του και εισηγητού. Επόμενος ο μιλητής, η κυρία Βίρινγκ, εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Βεβαίω ε, θεωρούμε και εμεί ότι 120 εκατομμύρια για τον ορίζοντα Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην έρευνα και στην ε, καινοτομία ακριβώ για να εξυπηρετήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε και να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Το ΠΔΠ είναι ένα ολόκληρος προπολογισμό. Ε, αλλά δεν ε, πρέπει να μιλάμε μόνο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά αντικείμενα που αφορούν τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραέξω. Πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις ε, πρέπει επίσης να δούμε ότι αυτές λαμβάνονται στα ταμεία και όχι στο πι δελτα πι. Οπότε οι συγκεκριμένες ε, κινήσεις και αποφάσεις μπορούν να ληφθούν στο επίπεδο των ε, ταμείων. Αυτά από μένα ως μια σύντομη εισαγωγή. Ευχαριστώ. Thank you very much, madam. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σακοράφα, εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ενδιάμεση έκθεση και τη θέση του Κοινοβουλίου ενώπιση της Συμφωνίας. Η γνωμοδότηση, κατά την άποψή μου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να σημειώσω εδώ την, τα σημεία συνένεσης που, και, διαφωνίας που μπορώ να έχω απέναντι σε αυτή την έκθεση. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι η νέα προγραμματική περίοδος να μην αποτελέσει, όπως και η προηγούμενη, προϊόν μια ταραχώδους διαπραγμάτευσης. Είναι ο καθήκον μας όλων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο να φροντίσουμε ώστε η διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί έγκαιρα και να μην καταλήψει σε χαμηλότερο όριο συνολικών δαπανών σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Η προτινόμενη συνολική αύξηση του προπολογισμού τη νέα περίοδου εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, είναι δειλή και υπολείπεται το σύνθετο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θεωρώ ότι ο αναδιανεματικός και επενδυτικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ικανότητα αντίδρασής της δεν μπορούν να εξασφαλιστούν αν ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 δεν οριστεί στο 1,3% ελάχιστον του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος γιατί όσο πιο μικρό σε μέγεθο και φιλοδοξία είναι ο προπολογισμό, τόσο πιο αναποτελεσματική θα αποδειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στου στόχου που έχει βάλει και στο ρόλο που θέλει να διαδραματίσει. Δεύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθέτης και δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο δικαιούται και πρέπει να έχει πλήρη και πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, της διαπραγματεύση, τη έγκριση εφαρμογή αξιολόγησης, ελέγχου και ολοκλήρωσης της νέας προγραμματικής περίοδου. Κάθε προσπάθεια παραγωνισμού, το κατά την άποψή μου, αποτελεί πλήγμα εναντίον του θεσμού και μεγαλώνει το, το, χάσμα όλο ένα και περισσότερο του δημοκρατικού ελλείμματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγηση <clears throat> της εφαρμογής της προγραμματικής περίοδου 21-27, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2023, η οποία θα συνοδεύεται από πρόταση για υποχρεωτική αναθεώρηση με συγκεκριμένη διαδικασία, με δεσμευτικές ημερομηνίε και με σεβασμό στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κλείνοντας την παραβασή μου, κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω ότι για μένα και την ομάδα μου, την QNGL, πρωταρχική σημασία έχει το ποιες πολιτικές επιλέγονται, εφαρμόζονται, ελέγχονται και αξιολογούνται για μας η επιλογή είναι μονόδρομος, γιατί επιλέγουμε να στηρίξουμε πολιτικές προς όφελος των πολιτών με στόχο την ανάπτυξη, την άρση των ανισοτήτων και την κοινωνική ευημερία, με όχημα τις δημόσιες επενδύσεις ικανές να καλύψουν το επενδυτικό χάσμα, με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία που υλοποιούνται με επιχορηγήσεις και επιμερισμένη διαχείριση, που προκαλούν συνέργειες και ε, εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα, μακριά από τις νεοφιλελεύθερες κατασκευές της οικονομικής διακυβέρνησης, της καταστροφικής λιτότητας και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, κλείνω κύριε Πρόεδρε, επιλέγουμε να στηρίξουμε πολιτικές για ειρηνικούς σκοπούς, μακριά από την στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε και στο πλαίσιο αυτού θα κινηθούν και οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την Thank you Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ο κύριος Σαουντάργας έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ε, σας υποστηρίζω και σας συγχαίρω για την έκθεση, εκτός από ένα σημείο. Δεν θα σας εκπλήξει. Ε, έχουμε 552 εκατομμύρια και χρειαζόμαστε 180 εκατομμύρια για την Ιγναλίνα. Γιατί αυτή τη στιγμή το project αυτό μπαίνει ε, σε μια επικίνδυνη φάση όπου θα αρχίσουμε να κλείνουμε ε, κάποιους ε, πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου Τσερνομπίλ. Είναι ένα μέρος της δουλειά που δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχω κάποιους υπολογισμού εδώ, βεβαίω δεν έχει νόημα να σας τα πω. Πριν από 20 χρόνια είχα μελετήσει αυτόν τον αντιδραστήρα ε, λεπτομερώς. Είχα συζητήσει με τον Επίτροπο Βαντεμπρούκ και είναι πραγματικά επικίνδυνος ο αντιδραστήρας αυτός. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, βασιζόμαστε στις ε, τροπολογίες σας για το θέμα αυτό έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Θα προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα γίνουν όλα δεκτά. Κατόπιν ο κύριος Ρουμπίχη. Είναι εδώ? Ωραία. Ναι, περιμένουμε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να υπογράφουμε κιόλας που και που γιατί βεβαίως ε, το χρήμα είναι κινητήριος ε, δύναμη και είναι σημαντικό το ότι είχα μια καλή έκθεση από τον Πασκάλ Λαμή και την ομάδα του ο οποίος μας είπε ότι έχουμε τρεις επιλογές. Ε, μία είναι να συνεχίσουμε όπως ήταν τα πράγματα ή να μπει ένα 50% στον προπολογισμό και θα έχουμε κάποια αύξηση αλλά η καλύτερη αύξηση για τις Δουλειέ και το ΑΕΠ θα είναι να διπλασιάσουμε το ποσό, δηλαδή 160 δισεκατομμύρια που απαιτούνται για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες μας. Οπότε στηρίζω τον φίλο μου τον Νίκ και χρειάζεται μια κόκκινη γραμμή και η κόκκινη γραμμή είναι τα 120 και οτιδήποτε παραπάνω από αυτό βεβαίως καλό είναι. Οπότε πρέπει νομίζω να κινηθούμε γρήγορα να έχουμε μια σαφή δέσμευση για τα 120 χωρίς καμία έκπτωση γιατί αυτά είναι απαραίτητα και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού αν χρειαζόμαστε κάτι για το στρατιωτικό, ναι εντάξει να τα δούμε αλλά θα πρέπει να αφαιρεθεί μετά από τα 120. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Και θα ήθελα τώρα στο επόμενο Βρίσκεται κάποιος εδώ από την ε, Επιτροπή. Ωραία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι εδώ. Εμείς απλώς βεβαίως σας ακούμε και αναμένουμε την έκθεση. Έτσι δεν έχω κάτι να προσθέσω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ ε, για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ γενικότερα για την υποστήριξη συνάδελφοι. Ε, βεβαίως υπάρχουν κάποια ζητήματα σημαντικά για εσά τα οποία θέλετε να προσθέσετε και είμαι έτοιμο να τα συζητήσω. Θα τα ψηφίσουμε αυτά. Ε, στις 9 Οκτωβρίου, όπως είπα, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών την 5η αυτής της εβδομάδας. Πολύ σημαντικό αυτό. Και θα φανούμε βεβαίω ευέλικτοι. Θα δούμε τι μπορούμε να υποστηρίξουμε ως Επιτροπή Ήτρε και θα δούμε ποια είναι και τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα επιμέρους τα οποία θα προσθέσετε εσείς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Όπως γνωρίζετε, είναι κρίσιμο το ζήτημα αυτό, όχι μόνο για την Επιτροπή Ήτρε, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη και το κανόνα συμμετοχής και διάδοσής του. Η συγκητής είναι ο συνάδελφος ο Νταν Νίκα. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα μαζί με το σημείο 5 της σημερινής διάταξης, πρόταση απόφασης ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Horizon Ευρώπη, εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος πλαισίου έρευνας και καινοτομίας, εδώ η συγκητής ο συνάδελφος Κρίστιαν Έλερ. Όπως ξέρετε, είναι ευθύνη δική μας τα προγράμματα πλαίσιο. Ανέκαθεν, είμαστε λοιπόν η Επιτροπή η οποία ηγείται των ζητημάτων αυτών και οι δύο εισηγητές έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης το συντομότερο δυνατόν, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θα θυμάστε ότι είχαν μόλις λίγες εβδομάδες να προετοιμάσουν το σχέδιο έκθεση λίγο πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι για να μπορέσει να υπάρξει έγκριση τώρα. Ήταν σημαντικό να ολοκληρωθούν και εργασίε μετάφραση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η προθεσμία τώρα για την υποβολή τροπολογιών ήταν η 6η Σεπτεμβρίου Η ανταλλαγή απόψεων λοιπόν αυτή είναι ε, μια δυνατότητα που δίνεται για να μπορέσουν οι συγκεκριτές να παρουσιάσουν πιο λεπτομερώς τις ε, απόψεις τους, τις προτάσεις τους και βεβαίως να συζητήσουν ε, και τα υπόλοιπα μέλη, της τροπολογίας που έχουν ήδη υποβάλει Έχουμε πάνω από 3.000 τροπολογίες, όπως γνωρίζετε, όπως πάντα βέβαια. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την ατζέντα έως τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι απαραίτητο για να ξεκινησουμε πραγματευσεις διαπραγματεύσεις Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ενδεχομένως ήδη και το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η πρώτη μας επιλογή. Θα δούμε εάν θα τα καταφέρουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Ο Ντάν Νίκα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, δεν ήταν εύκολο να εκπονήσουμε μία έκθεση για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπης. Ήταν ε, μία διαδικασία με πολλές προκλήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μπορέσαμε να διανύσουμε αυτό το σημαντικό στάδιο και ευχαριστώ τον Επίτροπο Μοέδας και τους διευθυντές Μπόρκες και Πάκες που ήρθαν σε μία διάσκεψη στο Βουκουρέστι και κάναμε και μία άλλη στις Βρυξέλλες. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολλές προτάσεις και μπορέσαμε να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δεν, ε, δεν λειτουργούσαν στο προηγούμενο πρόγραμμα και πρέπει να αλλάξουν. Τώρα, Horizon Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα απλό πρόγραμμα προσβάσιμο και να προωθεί μια συμμετοχή ισότιμη και διαφανή. Χαιρετίζεται το γεγονός ότι ο Horizon Ευρώπη διατηρεί τους τρεις πυλώνες, όπως το ορίζοντας 2020. Ο πυλώνας 2 και 3 όμως δεν περιγράφονται με σαφήνεια από την Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη, στον πυλώνα 2 έχουμε την έννοια των αποστολών, όμως το κείμενο παραμένει αρκετά όριστο. Το ίδιο ισχύει και για τον πυλώνα 3. Επίσης, το, Συμβούλιο της Ευρω... το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Καινοτομία με είναι ιδέα που τη χαιρετίζω. Θα πρέπει να περιγραφεί ε, με σαφήνεια. Οι δραστηριότητε του θα πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια γιατί δίνεται ένα σημαντικό κονδύλι του προπολογισμού η πολυπροκότητα και υπερβολικά πολλές ε, προτάσεις ε, ήταν ε, προβλήματα προσπάθησα να αντιμετωπίσω στην έκθεσή μου. Το πρόγραμμα Horizon 2020 είχαν κατατεθεί πάρα πολλές χιλιάδες αιτήσει τα κύρια σημεία του σχεδίου. Ένας πραγματικός προϋπολογισμός ε, και χαίρομαι που είχαμε την υποστήριξη όλων των σχεδόν εισογητών. Είχαμε τέσσερις συναντήσεις μέχρι τώρα, στο πλαίσιο των οποίων ε, συμμετείχαν και οι βουλευτές αλλά και οι βοηθοί και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε ως δυνατόν περισσότερες ιδέες που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να έχουμε μία έκθεση ικανοποιητική για όσο το δυνατόν ε, περισσότερους ε, συναδέλφους ε, αλλά και τους δικαιούχους. Έχουμε 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές στον προϋπολογισμό εγώ ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, για την υποστήριξη αυτή. Η βασική έρευνα και συνεργατική έρευνα θα πρέπει να και στηρίζει το πρόγραμμα όλα τα στάδια της καινοτομίας αλλά και τη βασική έρευνα και θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο και η έρευνα αριστείας. Το τρίτο, αμοιβαιότητα στις διεθνείς συμπράξεις γιατί θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ε, και η αρχή της αμοιβαιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά εκεί όπου είναι δυνατόν. Κατόπιν, τέσσερα, αυστηρότεροι κανόνε διανοητική ιδιοκτησία. Η έρευνα κοινοτομία συνδέονται άμεσα με τη διανοητική ιδιοκτησία. Χρειαζόμαστε σαφεί κανόνε σε αυτό το τομέα είναι ουσιαστικό για την προστιθέμενη αξία της έρευνας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ειδικότερα μικρότεροι και νέοι συμμετέχονται στο πρόγραμμα χρειάζονται συμβουλές ε, για τη διανοητική ιδιοκτησία προκειμένου να την προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο. 5. Αρχή τη πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άριστες ε, επιδόσεις σε ε, επιστημονικές δημοσιεύσεις, όμως όταν ε, μιλάμε για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αυτών, αυτά τα αποτελέσματα πολύ συχνά τα εκμεταλλεύονται συνήθω οι ανταγωνιστέ μα παγκοσμίω. Έτσι λοιπόν πρότεινα αυτή την ιδέα τη πρώτη εμπορική εκμετάλλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπο και η προσθέμενη αξία ε, των δαπανών που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, των φόρων που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, κατόπιν συνέργεια με άλλα ταμεία τη Ένωση για να ε, μειωθεί ο πολύπλοκο χαρακτήρα, ε, χρειάζεται να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των διάφορων μέσων χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και να, χρηματο... να χρησιμοποιηθούν ενιαίοι κανόνε και να έχουμε τη σφραγίδα αριστεία που θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο το πρόγραμμα. 7. Εγώ χαιρετίζω την εισαγωγή των αποστολών, όμως ε, θα πρέπει να οριστούν καλύτερα και θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, μετά από μια αρχή περίοδο, λαμβάνουμε σε υπόψη τη δικασία επιλογή και τη διακυβέρνηση. Πρέπει και το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στο σχεδιασμό των αποστολών. 8. Ίση αμοιβή για εργασία ίση αξία. Πιστεύω κράτοντα την αρχή τη ίση μεταχείριση και τη ίση αμοιβή ε, για εργασία ίση αξία στο πλαίσιο ενό ευρωπαϊκού προγράμματο που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλονται από το ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρέπει να υπολογίζονται με βάση ένα κοινό αλγόριθμο που καθορίζει τι επιλογέ του Ευρωπαϊκού Συγητή στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ενιαία κλίμακα που ισχύει για όλου του ερευνητέ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγή του ερευνητή, την τοποθεσία του ερευνητικού οργανισμού. Αυτή η μοναδική κλίμακα θα μπορούσε να βασίζεται στα επίπεδα σταδιοδρομία των ερευνητών, όπω ορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις σταδιοδρομίες στην έρευνα 9 ε, η ανώνυμη αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από εξάρτητου εμπειρογνώμονε. Είναι σημαντικό τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι δικαιούχοι να εμπιστεύονται το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Έτσι λοιπόν προτείνω ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε να προβαίνουν σε ανώνυμη αξιολόγηση των προτάσεων. Αυτό θα διασφαλίσει μια αμερόληπτη αξιολόγηση των προτάσεων που θα λαμβάνει υπόψη την προστέμενη αξία των έργων και κριτηριστία. Θα εκαπλούστευση Έχουμε την αξιολόγηση σε δύο στάδια, εσωτερική αξιολόγηση, αμοιβή εμπιστοσύνη ελέγχου και αποδοχή των συνήθων λογιστικών αρχών των δικαιούχων. Για περαιτέρω απλούστευση, προτείνουμε την εφαρμογή ενιαίων ποσοστών χρηματοδότησης σε ολόκληρο το πρόγραμμα. 11. Διεύρυνση προκειμένου η να μεγιστοποιήσει το δυναμικό τη έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να ξεπλώσει την αριστεία πιο ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να αντικοπτεριστεί και σε ποσοστά απορρόφηση. Έχουμε τώρα 87,2 εκατομμύρια της ολικής χρηματοδότησης, ενώ ε, η Ευρώπη 13, 4 και οι συνόμενες χώρες, 7% της συνολική χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ε, ενίσχυση της ελκυστικότητας ε, της Ένωσης. Τελική επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από το πόσο μπορεί να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονε και επιχειρήσει για να διεξαγάγουν έρευνα και να επενδύσουν στην Ένωση. Επομένως, ε, τα σχέδια που προσελκύουν άριστου επιστήμονε και επιχειρήσει από τρίτες χώρε θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετο οικονομικό κίνητρο. Και κάτι για το Brexit. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σε μία μοναδική ε, κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κρατός μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τώρα. Δεν υπάρχει καμία παράγραφος ε, όπου να μπορεί να ενταχθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 28, το 28ο κρατών μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε μεταβολή θα προέρθει από, από διαπραγματεύσεις μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και δεν βλέπουμε τίποτα στην έκθεση αυτή. Έτσι λοιπόν θέλω να αναφέρω ότι αυτό που ε, αναφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, παίρνουμε το σχάρι, θα θεωρηθεί ε, το Ηνωμένο Βασίλειο σαν τη Νέα Ζηλανδία ή σαν τον Καναδά. Δεν υπάρχει καμία όμως τέτοια αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή ήταν η σύντομη παρουσίαση, Πρόεδρε. Θέλω να του ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου και την Κομισιόν για την υποστήριξη που μου έδωσαν σε μια πάρα πολύ σύντομη περίοδο να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την έκθεση. Uh, uh, Τώρα θα ήθελα να δώσουμε λόγο στους κύριους εισηγητές. Α, συγγνώμη. Βεβαίως, ναι. Ο κύριος Έλερα αλλά όχι ως σκιώδης εισηγητής, αλλά ως εισηγητής για το δικό μας ε, το πρόγραμμα που εφαρμόζει τον ορίζοντα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με κάτι διαδικαστικό. Θα μάθατε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε αντίθεση με τα όσα μας είχε πει το Συμβούλιο στην αρχή, ε, για το το Συμβούλιο αμφισβήτησε την συναπόφαση στο πρόγραμμα αυτό, γιατί έχουμε άρα ένα πρόβλημα τώρα εδώ, Τι έχουμε το γενικότερο και το ειδικότερο πρόγραμμα που αφορά την εφαρμογή κομισιών, αποφάσισε να τα χωρίσει αυτά. Τώρα έχουμε λοιπόν δύο εκθέσεις με τους ε, κανόνες να αφορούν εν μέρη το ειδικότερο πρόγραμμα και εν μέρη την κυρία έκθεση και δεν υπάρχει λόγος να το αμφισβητήσει το Συμβουλίο και χαίρομαι για το ότι η Κομισιόν επιμένει στην νομική της θέση αλλά όλα τα επιχειρήματα που είχαν ακουστεί νομίζω είναι ιδιαίτερως προβληματικά γιατί δείχνουν ότι το Συμβούλιο προφανώς δεν θέλει να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία και εάν αρχίσουμε τώρα να μπλέκουμε σε διοργανικούς ε, καυγάδες ε, δεν είναι και πολύ κολακευτική εικόνα για μια Ευρώπη η οποία υποτίθεται ότι αντιλαμβάνεται ότι η καινοτομία είναι σημαντική για τις δουλειές και την ανάπτυξη και γενικότερα σε καιρούς ε, δύσκολους όπου αμφισβητείται και η ελευθερία της έρευνας στη ΣΥΠΑ για να μην πω για Κίνα, Ρωσία κτλ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ελευθερία της έρευνας και να μην περάσει τώρα σε αυτό το θέατρο σκιών για τις αρμοδιότητες. Τώρα, το τον λεχθέντο νομίζω πως υπάρχει μια κοινή ε, συμφωνία για το ότι το πρόγραμμα το ειδικό θα πρέπει να διαχωριστεί το θέμα της άμυνας για νομικούς λόγους και πρέπει να επιμένουμε σε αυτόν τον διαχωρισμό. Δεύτερον, υπάρχει επίσης μια συμφωνία και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου πάντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι θετικό το ότι και οι δύο εισηγητέ ε, δείξαν ακριβώς την διάθεση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για ζητήματα επίσης ε, μοναδικών δικαιούχων και για κάτι άλλο το οποίο επίσης μας ανησυχεί. Το Κοινοβούλιο, ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο ανέλαβαν την πρωτοβουλία και ε, όσον αφορά τις προτάσεις των εισηγητών για τα κονδύλια, τον διπλασιασμό του προπολογισμού και το πώς ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι εάν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να γίνει μόνο με το πρόγραμμα έρευνα. Το πρόγραμμα έρευνα αφορά την αριστεία, υπάρχουν κάποια όρια και πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους μας ε, και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν έχει νόημα να έχουμε μία νέα έκφραση λεγόμενη αυτή σφραγίδα της αριστείας ε, και να λέμε ότι κάποια είναι πάρα πολύ καλή αλλά δεν έχουμε κονδύλια. Μετά να τους χρηματοδοτήσουμε από τα διαρθρωτικά ταμεία όπου τους παραπέμπουμε. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών προγραμμάτων και των διαρθρωτικών ταμείων, αλλιώς δεν έχουμε και κάποιο ε, μοχλό πίεσης. Και αυτό το οποίο πρέπει να ξαναδούμε είναι το θέμα της ε, διεθνοποίησης. Συμφωνώ με τις ε, ανησυχίες της ε, Ντανίκας ότι πρέπει να το ξαναδούμε, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το ΕΛΚ θεωρούμε ότι πρέπει να αποφύγουμε οτιδήποτε το οποίο μπορεί να δείξει ότι η Ευρώπη πηγαίνει σε μια κατεύθυνση πρώτα η Ευρώπη πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και αυτό είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και ε, τη στιγμή που η Κίνα γίνεται πιο εθνικιστική, η Ρωσία επίσης, έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που λέει ότι η κλιματική έρευνα δεν είναι έρευνα αλλά είναι βουντού. Ε, πρέπει λοιπόν ο ρόλος της Ευρώπης να είναι ότι θα είμαστε εμείς το μέρος εκείνο του κόσμου που θα είναι ανοιχτό και δεν θα καθορίζουμε τα πάντα από τη δική μας την σκοπιά, γιατί βεβαίω η, κλιματική έρευνα είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Βεβαίως, εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά στο πώς ξοδεύουμε τα λεφτά Αλλά εάν υπάρχουν, αν δοθεί κάπου αλλού στον κόσμο μια επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο έρευνα. Ε, δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα, η πρόταση της Κομισιόν για να ξαναδούμε το ζήτημα για να υπάρξει και επαφή με την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους είναι σωστό, αλλά τελικά θα πρέπει να υπάρξει μια πράξη καταξιοδότηση. Δεν είναι κάτι το εξωτικό, όπως το θεωρεί το Συμβούλιο, για τις αποστολές πρέπει να έχουμε νομίζω κάποια ε, διοικητικά συμβούλια κάπως πιο διαφορετικά, να τα ξαναδούμε μετά από δύο χρόνια. Για τις συνεργασίες ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αναφέρονται στο ότι θα πρέπει ακριβώς ε, να δούμε την συνέχεια που θα πρέπει να υπάρχει και να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των εισφορών σε χρήμα και σε είδος και να περιοριστεί επίσης η χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από την διαδικασία διαβούλευσης, αλλά τελικά πρέπει να είναι πράξη κατεξοδότηση. Για τον δημιουργικό κλάδο αυτό είναι κάτι το καινούριο, νομίζω είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου γιατί είναι ένας παράγων πολύ σημαντικός για την οικονομία της Ευρώπης και για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ε, μας λένε ότι η δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει μια κινητήρια δύναμη για το μέλλον. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα νομίζω πω είναι κάτι το ταμπού ας πούμε, αλλά εντάξει πρέπει να δούμε λίγο τα proof of concept τώρα για για το φύλλο δεν αρκεί να το αναφέρουμε μόνο 182 φορές. Παραδείγματο χάρη στην επιχορήγηση Marie Curie θα πρέπει να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Να αναφέρουμε κάτι συγκεκριμένο για το εάν αλλάζει η οικογενειακή κατάσταση, όχι μόνο να λέμε 182 φορές τη λέξη φύλλο. Για ε, το fast track νομίζω πράγματι γεγονό είναι ότι μπορεί να είναι πολύ αργό το ερευνητικό πρόγραμμα, οπότε υπάρχει ένα νέο καινοτόμο μέσο εδώ για την διεύρυνση είπα ήδη κάτι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Και έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων στόχων και των αναγκών και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής βεβαίως το εάν θα έχουμε επιχορήγηση, δάνεια και εγγυήσει είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί και η διαδικασία αξιολόγησης είναι πάρα πολύ άργη για να μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε κάποιες καινοτόμες διαδικασίες και κάποιους δείκτες, δηλαδή εάν χρειάζεται να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά καινούριο πρέπει να υπάρχει και μια πολύ γρήγορη αξιολόγηση και ευελιξία. Πράγμα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είναι και αυτό ένα ζήτημα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε επίσης να προσελκύσουμε κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου στα σχετικά έργα. Και να αναφέρω κάποια ζητήματα. Πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό νέφος ε, επιστημών, το συζητάμε εδώ και 10 χρόνια, και τον ανάλογο προπολογισμό και ένα στόχο χρονικό. Για τα κλάστερ. αυτά για την ενέργεια. Πραγματικά κοιτάμε να δούμε πώ θα στηρίξουμε τα μέσα εφαρμογή για τι πράσινε λύσει στην βιομηχανία, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργεια, αλλά για την εφαρμογή στην βιομηχανία. Ένα νέο τομέα παρέμβαση για να εστιάσουμε στις βιομηχανικέ εγκαταστάσει γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να προσαρμοστεί. Θέλουμε επίση να έχουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την ασφάλεια. Δεν έχει νόημα να τα βάλουμε όλα μαζί Και πρέπει να υπάρχει επίσης και ένα εύρωστο πρόγραμμα για το δημιουργικό κλάδο, για την υγεία επίσης ε, εδώ και χρόνια ζητάμε να υπάρχει ένα επιστημονικό συμβούλιο για να συντονιστούμε σε θέματα υγείας. Έχουμε 1.800 τροπολογίες και ε, αρκετές εκατοντάδες έγραψαν και οι συγητές. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα αλλά και να αντιληφθούμε και να δώσουμε στο Συμβούλιο να καταλάβει ότι υπάρχουν τρόποι να το, να το καθυστερήσουμε, να το κάνουμε πολύπλοκο. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού στο... στην ε, κβαντομηχανική έχουμε κάποιες προόδους, ε, είμαστε σε ορισμένους τομείς πιο μπροστά από τους Αμερικανούς. Αν να περιμένουμε μέχρι το 2020 θα χαθεί η πρόοδος αυτή Πρέπει να κινηθούμε λίγο γρήγορα. Είναι και αυτό το νόημα της χειροτομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεπέρασα τα 10 λεπτά, αλλά ο συνάδελφο Έλερ ε, μιλούσε εδώ με διπλή ιδιότητα ως εισηγητής και ως κοιόδης εισηγητής και για το βασικό πρόγραμμα. Ο συνάδελφο Ζωρίνιο τώρα, ο οποίο ε, αντικαθιστά την κυρία Καμπεθόν Ρουίθ, έχει μόνο μία ιδιότητα, ε, ως σκιώδης εισηγήτρια ε, σε συγκεκριμένα επιμέρους προγράμματα. Κύριε Θωρίου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρεται η κυρία Καμπεσορουής, δεν μπορεί να είναι παρούσα. Εγώ θα παρουσιάσω τα κυρία σχολιά της, με τα οποία συμφωνώ και εγώ. Έχω συνυπογράψει πολλές από τις τροπολογίες και στις δύο εκθέσεις. Καταρχήν θέλω να Συγχαρώ τους δύο συγγητές, Δανικά και Κρίστιαν Έλερ, για τις εξαιρετικές εκθέσεις που έγιναν μέσα σε μια πολύ μεγάλη πίεση χρόνου. Όμως μας επιτρέπουν να έχουμε μια βάση εργασίας, ένα πρόγραμμα θεμελιώδες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα θα έλεγα και για το μέλλον του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της κοινωνικής αλλαγής. Καταρχήν, Θέλουμε να τονίσουμε την εξαιρετική ισορροπία ε, των διάφορων συμφερόντων που διακυβεύονται. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ε, κινητοποιεί πολλούς stakeholders ε, και θέλει να δώσει το μέγιστο δυνατό όφελος στην κοινωνία. Υπάρχει η ιδέα να τεθεί η επιστήμη στην υπηρεσία της κοινωνίας και να υπάρχει πραγματική ε, δημόσια απόδοση των επενδύσεων και ο άνθρωπος τίθεται στο επίκεντρο των αποτελεσμάτων που θέλουμε να πετύχουμε. Προφανώς ε, έχει νόημα η αύξηση στα 120 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού, καθώς εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις αναπτύσσεται η έννοια της ανοιχτή πρόσβασης και της ανοιχτή επιστήμης και αυτά συσχετίζονται με ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αυτή την εβδομάδα το θέμα του copyright ε, και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τη γνώση η αριστεία ως κριτήριο αξιολόγησης να μην ε, έχει περιορισμούς, ε, αλλά να έχει τη συμμετοχή και την απλούστευση και όχι τον αποκλεισμό. Η πρόθεση και η κινητοποίηση των νέων ερευνητών και καινοτόμων στην αναζήτηση ταλέντων, ο σεβασμός για την ε, ισότητα των δύο φύλων, Θέλω να υπογραμμιστούν οι θεμελιώδεις συνέργειες μεταξύ του Ορίζον Ευρώπη και των περιφερειακών ταμείων. Η προσπάθεια της ε, μείωσης των ισοτήτων μεταξύ των ε, λιγότερων αναπτυγμένων και των περισσότερων αναπτυγμένων περιοχών, κάτι που θέτει προβλήματα στην επιλογή των προτάσεων, το θέμα του να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες, να επιληθούν τα προβλήματα και να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Το χάρη, το επίκεντρο στην υγεία προτείνεται από τη συναδελφό μου, ε, η έρευνα για τον καρκίνο, ε, για τις καρδιογκιακές νόσους και επίσης ε, τονίζεται και η σημασία της γαλάζιας οικονομίας. Το ορίζον Ευρώπη θα πρέπει να σχετίζεται πάρα πολύ με αυτά τα προγράμματα, όμως εμείς ε, θα ψηφίσουμε και το Connecting Innovator Facility, ένα μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης ε, για να δημιουργήσουμε ε, συνδέσεις στην Ευρώπη, το πρόγραμμα EU Invest, ακριβώς για να έχουμε κεφάλαιο για την εξέβρεση λύσεων. Όλα αυτά τα προβλήματα, τα προγράμματα πρέπει να λειτουργούν ολοκληρωμένα. Δεν πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ ανταγωνιστικότητα σύγκληση και συνοχή, γιατί όσο περισσότερη συνοχή έχουμε, τόσο περισσότερη ανταγωνιστικότητα έχουμε και όσο περισσότερη ανταγωνιστικότητα υπάρχει, τόσο μεγαλύτερη συνοχή. Και Φυσικά αυτό σχετίζεται με το ότι θα είμαστε πιο ικανοί να απαντήσουμε στις ανάγκε του πληθυσμού. Είμαι βεβαίω ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η πρόκληση. Όμως εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δείχνει τη στρατηγική σημασία που έχει το Horizon Ευρώπη για το μέλλον μας. Και χαιρετίζω και εκ νέου την εργασία των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ζουντανόφσκι θα πάρει το λόγο τώρα και θα μιλήσει εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ κύριος Κρασνοντιώσκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πραγματικά ειλικρινά να συγχαρώ τους εισηγητές οι οποίοι ήταν υπό πολύ μεγάλη πίεση, χρονική. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής ε, και για τα δύο έγγραφα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω εν συντομία ποια σημεία πρέπει να υποστηριχθούν και ποια χρήζουν διευκρινήσεων. Τα 120 δις καταρχήν, για να μην υπάρχει έλλειψη ισορροπίας. Ε, βεβαίως η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμη τομής για να πετύχει η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική παγκοσμίω. Σε ό,τι αφορά την ε, ίση πληρωμή, ε, εμείς συμφωνούμε με αυτό, διότι όποτε έχουμε ακολουθήσει διαφοροποιημένη ε, προσέγγιση, αυτό οδήγησε σε πολύ δυσάρεστες συζητήσεις ε, ε, και αντιπαραθέσει στις ομάδες των ερευνητών και όπως είπε ο συνάδελφος ο κ. Νίκα πρέπει να βρεθεί μία ενιαία προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση και σε ό,τι αφορά τι αμοιβέ για να μην δημιουργείται ουσιαστικά φθόνος σε ό,τι αφορά το widening ε, έχει σημασία η αριστεία βεβαίως για την ε, επιστημονική δουλειά. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ισορροπίας έτσι όπως θεσπίστηκαν τα προγράμματα αυτά. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε ε, να είναι πιο ε, αιτιολογημένη η σύνθεση των ομάδων ερευνητών. Η θέση του Βασιλείου βεβαίω είναι δύσκολο να την καθορίσει κανείς. Διαπραγματεύσει συνεχίζονται. Δεν γνωρίζουμε ε, σε ποια κατηγορία θα πρέπει να μπουν οι Βρετανοί, διότι για μας το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως ειδική περίπτωση. Σε σχέση, δεν είναι, δεν είναι την Νότια Κορέα, το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, ε, και η σημασία αυτής της μακροχρόνιας ε, συνεργασίας με τον Ηνωμένο Βασίλειο χρήζει ε, μιας λύσης ισορροπημένης για την συνεργασία μας. Ε, όχι, αυτό είναι υποφελές και για τον Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για μας. Μιλάμε για επιστημονικά προγράμματα όπου θα είναι απαραίτητο στα πλαίσια των συζητήσεων ε, για το Brexit να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Κριστιαν, ο προηγουμένως, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ρητά την ε, διαστημική έρευνα, διότι έχει μπει εκεί κάπου ανάμεσα στη βιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες. Ε, εγώ πιστεύω ότι η διαστημική έρευνα είναι ένα τόσο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρεται ρητά για να μην βρεθεί πιο χαμηλά από τη θέση που ε, της αρμόζει. Έχουμε ε, κάποιες τροπολογίες για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. Ε, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να παίξει ένα νέο ρόλο, να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ενέργειας. πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι κρίσιμα για το σύνολο της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό το οποίο χρειαζόμαστε. Είναι λοιπόν σημαντικό σε αυτόν τον πυλώνα να, ε, να καθορίσουμε τι θα συμβεί με τις περιοχές ε, που χρησιμοποιούν τον άνθρακα ή που παράγουν άνθρακα. Ε, πάντως ευχαριστώ και για μια φορά τους συναδέλφους που μπόρεσαν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να βρουν... Madame Biering. Ευχαριστώ από την Άλντε τώρα από του φιλελεύθερου ε, Έχει το λόγο η κυρία Βίρινγκ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκα και τον κύριο Έλερ για τη σκληρή δουλειά του σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αναμένω με μονησία τη συζήτηση και των 3.500 τροπολογιών με του συναδέλφου και πραγματικά ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε μια συμβαστική λύση τον Νοέμβριο. Στη δική μου πολιτική ομάδα ξεκίνησε η συζήτηση με τον εξή στόχο. Αριστεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να, το πετύχουμε αυτό μόνο επενδύοντα σε ε, άριστα project ε, για τη βιομηχανία μας ε, και για τις ε, νέες τεχνολογίες. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν αποκλήσεις από χώρα σε χώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Πρέπει να τις δεχτούμε και πρέπει να φανούμε δημιουργικοί στις λύσεις που θα βρούμε. Έχω όμως μια διαφορετική άποψη σχέση με τον κύριο Νίκα. Στου φιλελεύθερους εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι υποφελέ να δημιουργούμε υποκατηγορίες σε ό,τι αφορά την αριστεία. Θέλουμε περισσότερες ευκαιρίες για να βρεθούν συνέργειε μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε ως στόχο 3% επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία στο κάθε κράτος μέλος με βάση στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ στα ζητήματα όπου θα ήθελα να ζητήσω κάποιε διευκρινήσει από του συναδέλφου στου επόμενου μήνε. Θα πρέπει να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για την κατανομή του προπολογισμού και το συνολικό ε, στόχο των 180 δισεκατομμυρίων. Ο Horizon 2020 ε, ε, ακολούθησε μια διαδικασία απλοποίησης που στέθηκε από επιτυχία. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και υποστηρίζουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάμε προς μια εξέλιξη. Μια εξέλιξη ομαλή, όχι μια επανάσταση ριζική. Δεν πρέπει βεβαίως ταυτόχρονα να μην αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η αντιμικροβιακή αντίσταση, ε, τα πλαστικά τα οποία πρέπει να κλείσουν από τους ωκεανούς, ε, τεχνητή νοημοσύνη και αντίκτυπο στην κοινωνία ε, κβαντική μηχανική, οι υπερυπολογιστέ. Πρέπει να κάνουν τι σωστέ επιλογέ έτσι ώστε τα άριστα project να έχουν προτεραιότητα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι το πρόγραμμα πρέπει να μπει σε μια βάση πραγματική. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ε, σε ό,τι αφορά το τι αναμένουμε. Ή μάλλον, συγγνώμη, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γνωρίζουμε τι αναμένουμε από το στρατηγικό σχεδιασμό. Ως Ευρωβουλευτής χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω πιο ενεργά σε αυτό το πρόγραμμα χάρη στις πράξεις κατεξιοδότηση. Όμως, ελπίζω ότι αυτό δεν θα επιβραδύνει τη διαδικασία. Οι πιο σημαντικοί εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτά τα πλαίσια ε, είναι οι ερευνητές, η βιομηχανία, η, τα πανεπιστήμια, οι καινοτόμοι φορείς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια για αυτούς και ότι η διαδικασία θα μπορέσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις αγορές αλλά και στα εργαστήρια. Συμφωνώ με τον κύριο Έλε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σημείο ισορροπία μεταξύ έρευνα και καινοτομία ε, στο σύνολο του οριζόντα, στο οριζόντα Ευρώπη. Βλέπω πολλέ πολλές ευκαιρίες ό,τι αφορά ε, την ευρωπαϊκή καινοτομία, όμως ε, η αύξηση του προπολογισμού αφορά κυρίως τον τρίτο πυλώνα. Δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία χωρίς έρευνα. για να συνεχιστεί η καινοτομία θα πρέπει να επενδύσουμε για στην βασική έρευνα για να μπορέσουμε να δρέψουμε το ωφέλη στη συνέχεια. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές. Και γι' αυτό εγώ υποστηρίζω αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε για τα σχόλιά σου. Εκ μέρους τώρα των Πρασίνων, ο κύριος Νταλούντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα για τη βιωσιμότητα. Ε, τα προγράμματα έρευνα και καινοτομία χρειάζονται μια σαφή διάσταση για να αφορά το περιβάλλον. Οι επενδύσει στην τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία ε, είναι πολύ σημαντικέ ε, το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το καλοκαίρι ήδη είχαμε μια πρώτη γεύση από τις επιπτώσεις ε, της αλλαγής του κλίματος στην Ευρώπη με καύσονες, ε, ε, πυρκαγιές, πλημμύρες είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και χρονικά. Πρέπει από το εργαστήριο να μπορούμε να φτάσουμε στην αγορά γρήγορα και να, να φτάσουμε σε μεγάλε κλίμακε σε, σε καινοτόμε λύσει για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τη Συμφωνία του Παρισίου. Έτσι, λοιπόν, έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίε για την αύξηση του earmarking για το κλίμα σημαντικά. Θέλουμε επίση ένα σύστημα ευοπτεία το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να διαφανεί μηχανισμό που θα ε, εξασφαλίζει ότι η Κομισιόν θα πετυχαίνει του στόχου στο πρόγραμμα αυτό είμαστε πίσω κατά 5% σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, το στόχο για το, για το περιβάλλον. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Η Κομισιόν, το Ελληνικό Συνέδριο, αλλά δεν γίνεται τίποτα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το κενό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, πρέπει η ακυρεότητα τη αριστείας να παραμείνει δυσκολευόμαστε να δεχτούμε συμβιβασμού ό,τι αφορά το κριτήριο αριστεία. Διότι είναι το πιο, πιο σημαντικό συστατικό έτσι ώστε τα προγράμματα έρευνα και καινοτομία να είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα κενό καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να το καλύψουμε έχουμε πολλά και διάφορα εργαλεία στη διάθεσή μα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο όμω το κατάλληλο στην κάθε περίπτωση. Συνέργεια με άλλα προγράμματα, με του πολιτικού στόχου είναι ο πιο καλό τρόπο να πετύχουμε αριστεία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, θέλουμε ένα ανοιχτό πρόγραμμα ε, απέναντι στον κόσμο. Υπάρχουν λαϊκισμοί, υπάρχει, υπάρχουν φωνές απομονωτισμού, απομονωτισμού εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, όμως ε, μια Ευρώπη η οποία δεν θέλουμε να είναι μόνο για την Ευρώπη, να είναι μεγάλη μόνο για την Ευρώπη. Θέλουμε ε, ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα τη καινοτομία για όλο τον κόσμο. Επίση, στρατηγικό σχεδιασμό. Ω θεσμικό όργανο, θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και σχετική διαδικασία. Δεν μπορούμε να δώσουμε τι εξουσίε αυτέ αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιλέγει ε, το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, αλλά να έχουμε λόγο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τι στρατηγικέ προτεραιότητε του προγράμματο εργασιών. Αναμένουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με του συναδέλφου ε, σε ό,τι αφορά τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ε, Σα ευχαριστώ. Η Γκουε εκπροσωπείται από δύο μιλητέ, τον κύριο Σιλικιώτη σκιώδη συγητή για το πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για το πρόγραμμα που ετοίμασε ο συνάδελφο στο σχέδιο συγητής είναι ο Ντανίκα και η συνάδελφος η Μαρίσα για την έκθεση που η είναι ο, ο συνάδελφος ο Ε, πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντανίκα για την έκθεση που έχει ετοιμάσει αλλά ιδιαίτερα για την παραγωγική συνεργασία που επιδιώκει να έχει μόνο στις πολιτικέ ομάδες ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Η ομάδα της gue ε βλέπει εν γέννη θετικά τις προτάσεις που κατάθεσε ο εισηγητή για την έκθεση Horizon Europe και για μας προτεραιότητα να στηριχτούν προγράμματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στι σύγχρονες ανάγκες τη κοινωνία ώστε να υπάρξουν κοινωνικά ωφέλη. Ζητάμε λοιπόν να δοθεί όθηση στην έρευνα που επιδιώκει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων, στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στην πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων. Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγηση, έχοντα τώρα και την εμπειρία του προγράμματο Ορίζοντα 2020, θα πρέπει να επιδιώξουμε βελτιώσει μεγαλύτερη διαφάνεια και δίκαια διαμορφωμένε ομάδε αξιολόγηση. Αναφέρθηκε και ο συνάδελφο Οντάν Νίκα για αυτό το θέμα. Επίση, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα μέτρα που πρέπει να ληφθεί ώστε να στηριχθούν έμπρακτα οι πολύ μικρέ και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να μπορέσουν να αναπτύξουν δραστηριότητε έρευνα και κοινοτομία και να συμμετέχουν ισότιμα στο πρόγραμμα αξιοποιώντα τι ευκαιρίε χρηματοδότηση. Στόχο πρέπει να είναι να καταπολεμήσουμε τι όποιε ανισότητε υπήρξαν μέχρι σήμερα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αλλά εξού σημαντικό είναι και να διασφαλίσουμε πως τα δεδομένα και οι γνώσεις που θα παράγονται από τα χρηματοδοτούμενα έργα θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Κλείνοντας, ε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικότερα και ειδικότερο θέμα και ευαίσθητο όπω είναι το θέμα τη υγεία. Είναι αδύρυτη ανάγκη να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Ορίζοντα Ευρώπη και να συνεχίσουμε το σχετικό κονδύλιο ώστε να προωθήσουμε την έρευνα στα βασικά θέματα υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τι σπάνιε ασθένειε, αλλά και τι χρόνιες ασθένειε. Η βελτίωση και η προστασία τη υγεία όλων των ανθρώπων με την άπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών θεραπείων για την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία για πλήρη ένταξη στην κοινωνία πρέπει να είναι κοινό στόχο όλων μα. Και πρέπει να πω ότι προ αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ματίας ε, για το ειδικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Έλερ. Εγώ αναφέρομαι στο ειδικό πρόγραμμα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Η βάση που παρουσιάστηκε εδώ αποτελεί καλή βάση εργασίας και υπάρχει πολύ κοινό περιθώριο. Τώρα, σε σχέση με κάποιες διαστάσεις που συζητήσαμε και στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά. Σε αυτά που θεωρώ απαραίτητα, ουσιαστικά. Αναφέρθηκε ήδη ο εισηγητής ότι δεν ε, υπάρχει ε, εύρωστη εστίαση σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Εγώ συμφωνώ, αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα. Γι' αυτό παρουσίασα την πρόταση να δημιουργηθεί ένα κλάστερ για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ε, ήδη εδώ και κάποιο καιρό που ε, φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να μειωθεί η σημασία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Όμω δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα πιο σημαντικό τομεί έρευνα στην Ευρώπη και πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα ε, στο να μείνει άθικτο αυτό ο κλάδο ε, και να ενισχυθεί μάλιστα. Γιατί. Ε, χρειαζόμαστε απαραίτητα τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες έτσι και χρειαζόμαστε και την ε, θεμελιώδη, τη βασική επιστήμη. Δεν υπάρχει καινοτομία χωρίς έρευνα και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη βασική έρευνα δεν ε, μπορούμε να μιλήσουμε ε, για ε, το ότι είναι νεκρές οι βασικές επιστήμες, γιατί αποτελούν τη βάση της καινοτομίας. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή της διάστασης της έρευνας και των βασικών επιστημών σε κλάστερ που υπάρχουν ήδη στο ίδιο το πρόγραμμα, στον τομέα της υγείας. Αυτό έχουμε μέσω της εισαγωγής σε αυτό το κλάστερ ενός ε, συνόλου τομέων έρευνας που έχουν παραλυφθεί, που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη ε, με τις ε, μη μολυσματικές ασθένειες, Παραδείγματο χάρη, αναφερόμαστε στο διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, σε σπάνιε νόσου. Αυτή είναι μια διάσταση που πρέπει να συμπεριλάβουμε. Όπω και οι κλιματικέ ε, ε, οι κλιματικέ αλλαγέ, η θαλάσσια έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί που δεν έχουν συμπεριληφθεί εδώ. Αυτή είναι η κυρία μου ανησυχία και θα κλείσω εδώ. Δεν υπάρχει καινοτομία χωρίς έρευνα και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτρέψει να έχουμε επιβράδυνση σε κάποιου από του πιο σημαντικού τομεί της έρευνας. Επομένως, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εγγυθεί την ε, πλήρη αμεροληψία για ανεξαρτησία ε, των ε, ερευνητών και απόλυτη διαφάνεια και αποσαφήνιση σε σχέση με τις ε, λειτουργίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του FTD, η κυρία Νταμάτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η αρχή speed over quality που έχει εφαρμοστεί με τις τροπολογίες ε, στον ορίζον Ευρώπης ε, για να προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν ε, την πρόταση της Κομισιόν πριν από τις ευρωεκλογές, δεν έχει αναδείξει το έργο μας και της Γραμματείας τις επόμενες εβδομάδες ε, θα έχουμε ε, κάποιες τροπολογίες ε, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θέλετε να ακουστεί μόνο η φωνή δύο ή τριών μεγάλων ομάδων, όμως η δημοκρατία πρέπει να είναι κάτι που το και για τις μικρές ομάδες. Βλέπουμε και μια διαδικασία διαδικασία του Συμβουλίου ε, να αφαιρέσει τις καθήκοντα του Κοινοβουλίου μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης πριν ε, δύο μήνες ε, είχε παρουσιαστεί η πρόταση του περιεχόμενο της απόφασης να ενταχθεί στον κανονισμό. Ε, όμως ε, σήμερα, ε, αν εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική, θα έχει ε, διευκολύνει πιο αποτελεσ... θα έχει διευκολύνει τη δική μας δουλειά και θα την έχει επιταχύνει. Όμως εδώ το μόνο που απομένει είναι να περασπίσουμε τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως είχε συμφωνηθεί. Θα συνεργαστούμε παράλληλα για να έχουμε ένα καλό συμβαστικό που θα βελτιώνει το πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της έρευνα και της καινοτομίας προς όφελο των πανεπιστημίων, των ερευνητών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η δική μας συνεισφορά στο πρόγραμμα πλαίσιο. Καταρχήν, ε, αφορούσε πέντε πτυχέ από διαφορετική σκοπιά διάφορες τροπολογίες δικές μας ε, αφορούν ε, την ε, τροπολογία του όρου κλάστερ έτσι όπως χρησιμοποιείται από την Κομισιόν. Ενώ για διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Γερμανία ο όρος είναι αμφίσιμος και ήδη χρησιμοποιείται για άλλα σχέδια. Κατόπιν, δώσαμε μια μεγάλη προσοχή στους στόχους που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδίως ε, στην επίτευξη του στόχους ε, μηδενικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και ζητούσαμε να αποκλείονται κατηγραμματικά κάθε είδος χρηματοδότησης και ενίσχυσης ε, στα ορυκτά καύσιμα. Η πρόταση της Κομισιόν κατόπιν δίνει έναν θεμελιώδη ρόλο ε, στην ε, ε, βιομηχανία και στην αγορά που φυσικά έχουν σχετικό ρόλο αλλά θα πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την αξία της έρευνας και στο κοινωνικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν εισαγάγει μια σωστή ισορροπία στο κείμενο δίνοντας, αποδίδοντας κατάλληλες προτεραιότητες και θετώντας ένα πλαίσιο που σέβεται περισσότερο τις αρχές που έχουμε στις συνθήκες της Ένωσης. Προσπαθήσαμε επίσης να δείξουμε ότι πρέπει να αποφεύγονται και δορσκοπικές πράξεις με τα διαθέσιμα κονδύλια, εκεί όπου ε, γίνεται προσφυγή σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, ε, έχουμε ε, ξαναεισάγει το εργαλείο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους εγγυόμαστε τη δυνατότητα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόσβαση των κονδυλίων για την έρευνα και την κοινοτομία. Αυτά είναι τα κυρία σημεία παρέμβαση που θέλουμε να υπογραμμίσουμε και ελπίζουμε να μπορούν να συνεισφέρουν σε βελτίωση του κειμένου της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Περνάμε στους άλλους μιλητές. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που σας βλέπω. Να ευχαριστήσω τον Ντάν και τον Κρίστιαν για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκαναν και πολύ λεπτομερή. Θα ήθελα όμως να επισημανώ ότι δεν είμαι ολόγραμμα. Ε, βρίσκομαι εδώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι ακόμα κράτος μέλος, νομικά και πολιτικά. Και Ντάν και Κρίστιαν, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας. Όπως λέτε Γέρζη συχνά στις διαπραγματεύσεις, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, δεν, μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη αλλάξει άποψη και αυτήν την στιγμή είμαστε κράτος μέλος. Καλώς ορίζω τις προτάσεις της Κομισιόν. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπαν ο Νταν και ο Κριστιαν, ειδικά όσον αφορά την αύξηση του προπολογισμού για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και την εστίαση στην απλοποίηση με βάση τις εμπειρίες εφαρμογής του ορίζοντα 2020. Επίσης, καλωσορίζω αυτά τα οποία ακούστηκαν για το φύλλο που λέει ο Ντάν ότι πρέπει να ενταχθεί επαρκώς στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά συμφωνώ και με αυτό το οποίο είπε ο Κριστιαν και άλλοι ομιλητές και ο Κάρλος για την ανάγκη τα κονδύλια αυτά όχι απλά να στέκονται, αλλά να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι ώστε ε, να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ίσως έχουν μείνει λίγο πίσω να μπορούν να έχουν ένα σκαλοπάτι για να φτάσουν στην αριστεία. Δεν μπορεί να αφήνουμε κόσμο να τον εγκαταλείπουμε. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την αριστεία στην έρευνα, της διεθνής συνεργασίας, να είμαστε ε, να έχουμε αυτές τις αρχές, ε, το να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και να ενισχύουμε την αριστεία. Κάποια σημεία πρέπει να περιληφθούν. Οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες ε, στο πλαίσιο της έρευνας που χρηματοδοτούμε επίσης πρέπει να περιληφθούν. Οπότε, Είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που έχει γίνει και για την συνένεση που υπάρχει και χαίρομαι και για την συνεργασία και την διαφάνεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δήλωσή σας και για την ε, δήλωση που κάνετε στην εισαγωγή σας. Και κατόπιν έχουμε τον κύριο Γκάιερ. Θα δοκιμάσω και πάλι την υπομονή σας φοβάμαι. Τέσσερα σημεία έχω να πω. Για τα ζητήματα εκπομπών και βιομηχανίας πρέπει να δούμε και την κοινωνία των πολιτών και ερευνητικών οργανώσεων. Επίσης, συμφωνώ με την ιδέα των πρασίνων ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να έχει κάποιες ε, μεγαλύτερη, να τη δοθεί μεγαλύτερο βάρος. Και πρέπει να υπάρχει κορυφαία έρευνα και να προσελκύσουμε κορυφαίους ερευνητές και τέλος, να επαναλάβω ακόμη μία φορά, πρέπει να φροντίσουμε ο ορίζοντας Ευρώπη να παραμείνει ε, πολιτικός και όχι στρατιωτικός. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, σας ευχαριστώ. Και τώρα έφτασε η στιγμή της Κομισιόν. Και του κυρίου Μπούτσερ. Αναπλέον του Διευθύντη της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας βέβαιως. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και ειδικά τους διευθυντές, τους κυρίους Ελερκένικα είναι την ευκαιρία που μου δίνουν να σχολιάσω τις ε, τροπολογίες. Ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει το μεγάλο σας ενδιαφέρον ε, και το ότι είστε προσιλωμένοι στο να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Μιλήσατε ε, για το θέμα της αρχήτητας και όπως είπε και ο πρόεδρος ελπίζουμε να καταφέρουν τα διαθεσμικά όργανα να επιτύχουν μια πολιτική συμφωνία για τον ορίζοντα Ευρώπη. Να σας πω κάποια πράγματα για την νομική βάση και μετά από κάποιες απόψεις για τις τροπολογίες για την νομική βάση. Όπως είπε και ο κύριος Έλερ, κάποια κράτη-μέλη ζήτησαν από το συμβούλ την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου να γνωμοδοτήσει για την νομική βάση του συγκεκριμένου προγράμματο και πράγματι η νομική υπηρεσία πρότεινε να φύγει το άρθρο 187.3 από την πρόταση τη Κομισιόν και όπω γνωρίζετε αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 182 παράγραφο 4 είναι η μόνη ενιαία νομική βάση. Θα μείνει η μόνη ενιαία νομική βάση. Θα φύγουμε από την τακτική νομοθετική διαδικασία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μόνο έναν συμβουλευτικό ρόλο. Οι συζητήσεις βεβαίως ακόμη γίνονται, όμως φαίνεται ότι κάποια κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν την θέση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, κυρίως επειδή το θέμα αυτό της νομικής βάσης θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο για άλλα προγράμματα. Όμως, Κομισιόν θεωρεί ότι η πρότασή της έχει νομική βάση και θα συνεχίσει να την υπερασπίζεται. Οπότε σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε ακριβώς να ζητάμε την τακτική νομοθετική διαδικασία. Για τον στρατηγικό σχεδιασμό, να θυμάστε ότι ο σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να προετοιμάσει το έδαφος για να συνταχθούν κάποια προγράμματα εργασίας και για τον ορίζοντα Ευρώπη θέλουμε ακριβώς να υπάρχει διαφανή και συνδημιουργία με άλλα θεσμικά όργανα και τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο να είναι ενήμερα πριν ξεκινήσει η Επιτροπολογία για το πρόγραμμα εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πρόθεσή μας είναι σωστή και προτείνουμε ακριβώ μια διαδικασία η οποία θα είναι ανοιχτή και σε συνεισφορές από τα άλλα θεσμικά όργανα και θα εγκριθεί τελικά από ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ο απλούστερο τρόπο για να έχουν όλε οι πλευρέ την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόσουμε τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές προτεραιότητες όπως επεσήμαναν οι βουλευτές. Με βάση αυτά, η Κομισιόν θεωρεί πως ε, οι πράξεις κατεξιοδότηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο, καθώς ο στρατηγικός σχεδιασμός ε, δεν έχει στόχο να συμπληρώσει το νομοθέτημα. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε αρκετή ευελιξία και να σεβόμαστε τα χρονοδιαγράμματα. Να μην ε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η εναλλακτική των πράξεων κατεφρομογή είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε για τους προϋπολογισμούς. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας ε, όσον αφορά τους προϋπολογισμούς για το νέο πρόγραμμα ε, είδαμε κάποιες τροπολογίες που προτείνουν σημαντική αύξηση για το κομμάτι της αριστείας ε, και μείωση για κάποια άλλα. Βεβαίως, εμείς ε, θεωρούμε πως η πρότασή μας είναι αρκετά ισορροπημένη μεταξύ των τριών πυλών και εντός αυτών, αλλά βεβαίως ευχαριστώ να ακούσουμε τα επιχειρήματά σας. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για να περιοριστεί η ευελιξία του υπερπολογισμού να μειωθεί από το 10% στο 5%. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω πως σε όλες τις προτάσεις του ΠΔΠ η Κομισιόν έχει πει ότι η ευελιξία είναι ένα μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από τα προηγούμενα χρόνια και θα θυμάστε οπωσδήποτε την κρίση έμπολα και ζήκα όπου είχαμε ακριβώ αυτήν την πολύ χρήσιμη ευελιξία. Το θέμα τώρα της ε, δομής ε, των κλάστερ αυτού του πυλώνα 2 ε, υπήρχε μια πρόταση να σπάσει σε ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν μια κοινωνία με ένταξη και ένα άλλο ασφαλής κοινωνία. Εμείς είπαμε να απομακρυνθούμε από την κεντρική ιδέα και να φύγουμε από την τομεακή καινοτομία και να πάμε στην συστημική καινοτομία. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια επιχειρήματα για να σπάσουν αυτά τα δύο κλάστερ, αλλά πράγματι θεωρούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να μας οδηγήσει σε μια κλαδική προσέγγιση και το βλέπουμε ήδη στο Συμβούλιο, όπου έχουν ακουστεί κάποιες ιδέες να πάμε από τα πέντε στα 8 κλάστερ. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όμως πλέον δεν θα μιλάμε για κλάστερ αλλά για κλάδους όπως και σήμερα. Οπότε θα απομακρυνθεί ε, έτσι η πρόταση αυτή από την αρχική ιδέα. Τώρα, για το χάσμα της καινοτομία συμφωνούμε τον στόχο να γεφυρωθεί αυτό και για τον λόγο αυτό προτείναμε τον προϋπολογισμό ακριβώς ε, της ε, αριστείας να διπλασιαστεί όμως ο στόχος του να γεφυρωθεί το χάσμα κατά 50% γύρει κάποια ερωτήματα όπως η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στόχων, το πώς μπορεί να μετρηθεί κάτι τέτοιο και πώς μπορεί ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων ε, να μετρηθεί χωριστά από τον αντίκτυπο εθνικών μέτρων. Είναι σαφές ότι η συμμετοχή ε, και άλλων χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική, οπότε κοιτάμε και ψηλές Παραδείγματο χάρη ε, κάποιες ε, υποτροφίες, ε, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου τις αρχές του αντικτύπου και της αριστείας που είναι τα θεμέλια του προγράμματος. Νέα κριτήρια για την κατάταξη των προτάσεων ίσως αποκλίνουν από αυτές. Επίσης θεωρούμε ότι μέρος της επιτυχίας του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι ακριβώς η επιμονή στην αριστεία. Τυχόν νέα κριτήρια θα την υπονομεύσουν. Η αξιολόγηση του συστήματος ε, αξιολόγησης δεν έχουν δείξει την ανάγκη κάποια τυφλής αξιολόγησης. Αλλά οι δυσκολίες αντιθέτως ε, πρέπει να συνεξεταστούν καθώς θα υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης νέων κριτηρίων επιλεξιμότητας, ανωνυμίας, αυξημένο διοικητικό κόστος και υψηλός κίνδυνος αποκλεισμού κάποιων προτάσεων και διάφοροι νομικοί κίνδυνοι. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και το θέμα των αξιολογιστών ως ποσοστό των νέων ερευνητών. Όσον αφορά κάποια εναρμονισμένα επίπεδα επιστροφής των ε, δαπανών θα πρέπει να πω ότι δεν πληρώνει ο ορίζοντας μισθούς σε ερευνητέ, αλλά αποδίδει το κόστος σε οργανισμούς. Οπότε η Εθνική φορείς έρευνας αποφασίζουν. Ε, αν έχετε την καλοσύνη, λέει ο Πρόεδρος, ε, λίγο πιο ανθρώπινα, γιατί δεν μπορούν να σας ακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ναι, λίγο πιο αργά παρακαλώ. Ναι, βεβαίω. Για την αρμονισμένη, τα αρμονισμένα επίπεδα αποζημίωση για όλου του ε, ερευνητέ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εμεί δεν πληρώνουμε μισθού στου ε, ε, ε ερευνητέ. Εμεί αποζημιώνουμε του ανθρώπου αυτού για το κόστο τη έρευνά του. Οι εργοδότε στα κράτη-μέλη είναι αυτοί που αποφασίζουν σε ό,τι αφορά του μισθού, τι αμοιβέ. Και δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει ε, μια ενιαία κλίμακα σε ό,τι αφορά τι αμοιβέ στον τομέα τη έρευνα ε, πανευρωπαϊκά. Βεβαίω είναι ένα θέμα που είναι ευαίσθητο και για μα. Η πρότασή μα λοιπόν προβλέπει να δεχθούμε ε, μόνο ποσά τα οποία ανταποκρίνονται στο ελάχιστο κόστο που προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο για τι αμοιβέ. Ε, το ε, προσωπικό κόστος ε, το μέσο για αυτούς που συμμετέχουν στο, στις υποτροφίες ορίζοντα 2020 είναι πολύ πιο υψηλό από το, το μέσο όρο σε κάθε χώρα με συγκρίσιμα στοιχεία. Ε, βεβαίως το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη θα πρέπει να μπει στο ευρύτερο τοπίο των προγραμμάτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζουμε τις ιδέες ε, για τη βελτίωση της συνέργειας. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της θέλει να συνεχίσει αυτό το άνοιγμα διεθνών συμμετοχών, διεθνής συνεργασίας ε, σε μια κλίμακα χωρίς προηγούμενο και θέλουμε να μπορεί να υπάρχει και ένα άνοιγμα προς τις συνδεδεμένες τρίτες χώρες, στο, στην, στην, καρδιά της στρατηγικής ε, της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της ε, καινοτομίας είναι τα κοινά συμφέροντα και τα αμοιβαία ωφέλη. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε να παραμείνει δυνατότητα για τους Ευρωπαίους ε, ερευνητέ να, να μπορούν να εργαστούν μαζί με τους καλύτερους ε, διεθνείς ερευνητές στον συγκεκριμένο κλάδο δεν πρέπει να νερώσουμε τα κίνητρα που έχουν οι χώρες που θέλουν να είναι συνδεδεμένες χώρες στα προγράμματα αυτά. Από την άλλη, και βεβαίως αυτό είναι πολύ σωστό, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες συμμετοχής προσφέρει κάποια εργαλεία ε, που προστατεύουν τα ειδικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών και των σχετικών οντοτήτων και σε ό,τι αφορά την μετάλλευση των αποτελεσμάτων. Για την EIC εμείς ε, χαιρόμαστε που υπάρχει υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, πιο καινοτόμες ε, και ριζικές λύσεις ό,τι αφορά την καινοτομία της. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την αύξηση της καινοτομίας. Θα πρέπει αυτά να καλύπτονται και από τον δεύτερο πυλώνα και από τα οικοσυστήματα έρευνας και τον πυλώνα 3 το σχετικό. Ε, είναι σημαντικό για το νομικό κείμενο να έχει αυτό το χαρακτήρα, να μην είναι ένα όχημα απλά για κάποιες γενικές πολιτικές ε, δηλώσεις. Σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις, ε, χαιρόμαστε που συμφωνείτε με τις κοινέ αποστολές. Ε, συγγνώμη, αλλά ούτε ο Επίτροπος δεν μιλάει τόση ώρα. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μα είπατε, λέει ο πρόεδρο. αλλά ολοκληρώστε, ολοκληρώστε, αν σα μένουν λίγα. Όχι, ήθελα απλώ να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξή σα ε, σε ό,τι αφορά τι αποστολέ και τι συμπράξει. Θα είναι καλό αυτό να καθορίζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ε, από του λόγου για του οποίου δεν υπάρχει προπολογισμό για τι αποστολέ ε, στην πρόταση, αξίζουν κάτι καλύτερο. Θα πρέπει πρώτα όμω να καθορίσουμε πώ θα εφαρμοστούν πριν επιλύσουμε ε, το θέμα τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ για του δύο εισηγητέ ε, για τι τις εκθέσει εκθέσεις για τι τροπολογίε και για την ευκαιρία που μου δώσατε να σα πω και εγώ τη δική μου άποψη για τα σχέδια τροπολογιών και συγγνώμη εάν αυτή την ευκαιρία εγώ την εκμεταλλεύτηκα σε υπερβολικό βαθμό. Μάλιστα, πολύ ευρεία η συζήτηση, τα σχόλιά σας ε, ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τους δύο εισηγητές ε, να συνοψίσουν τη συζήτηση, ε, τα σχόλια. Ο Νταν Νίκα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συνεισφέρω για τα σχόλιά σας από όλους ε, τους ε, σκιωδησηγητές και από όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Να πω μόνο ότι ακολουθεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη περίοδος. Θα πρέπει να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες και να εργαστούμε επί από, σε πάνω από 1.400 τροπολογίες. Και ο συνάδελφος Έλερα έχει λάβει 1.800. Πολύ έντονη περίοδος, δύο διευκρινήσεις μόνο σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έχουμε κάποιες νομικές απόψεις. Μου είπε το η υπηρεσία, η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να μην θίξουμε αυτό το θέμα, γιατί αυτό αφορά την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με το ΕΒ. Βασίλειο. Σε σχέση τώρα με το θέμα της αριστείας, δεν το εξηγήσαμε καλά. Τα υποκριτήρια αναφέρονται μόνο στην περίπτωση που δύο project ή περισσότερο έχουν ε, το ίδιο σκορ, δηλαδή αν έχουν ε, τις ίδιες επιδόσεις που τα διαφοροποίηση και έχουν εισαχθεί τα υπόλοιπα κριτήρια για να μπορούσαν να ε, να μπορούσε να γίνει επιλογή μεταξύ δύο project που έχουν τις ίδιες ε, επιδόσεις. Έχουμε πολλές φορές εξαιρετικά προγράμματα που παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνδεδεμένες χώρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο κύριος Έλερ. Τέλος, να μιλήσω λίγα γερμανικά. Κοιτάξτε. Όταν μιλάμε για 120 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι έχουμε αύξηση του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κάτω από τους στόχους του Συμβουλίου. Είχε πει το Συμβούλιο πριν από 10 χρόνια ένα 3% του ΑΕΠ, κάτι το οποίο θα σήμαινε 180 δισεκατομμύρια σήμερα. Γιατί κάθε χρόνο το Συμβούλιο επέλεξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρευνας για περικοπές. Οπότε, εντάξει, δεν είμαι καθολικός, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να δει ο καθένας εδώ πέρα τις ε, αμαρτίες που έχει κάνει. Αν λοιπόν δεν έχουμε έναν προπολογισμό 120 δισεκατομμυρίων, θα πρέπει κάποια να το πάρουμε απόφαση ότι θα χάσουμε το τρένο της καινοτομίας, το παγκόσμιο τρένο. Θα μας ξεπεράσει η Ασία, η Κίνα, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, στην Βόρεια Αμερική με έναν εξωτικό πρόεδρο, αλλά με έναν προϋπολογισμό ποσοτικά σαφώς και, και αναλογικά σαφώς υψηλότερο από την Ευρώπη. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι διατεθειμένος τώρα να συζητάω για την υποτιθεμένη αύξηση του, του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να επιμείνουμε στα νούμερα τα οποία έχει εγκρίνει ομόφωνα το Συμβούλιο. Και ένα νούμερο τέλος το οποίο είναι σημαντικό. 8 στις 10 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια βασίζονται στην καινοτομία. Η ιδέα στη δεκαετία του 90 ότι οι υπηρεσίες ε, θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας διαψεύτηκε. Δεν θα κοβεί ένα στα μαλλιά του άλλου. Πολύ απλά το κοινωνικό μας μοντέλο θα χρηματοδοτήσει στην Ευρώπη μόνο αν είμαστε αρκετά καινοτόμοι και είμαστε σε θέση να δημιουργούμε έτσι κάποια πράγματα, να έχουμε από εκεί φορολογικά έσοδα κτλ. κτλ. Και τέλος, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να δουν τις λεπτομέρειες ε, των τροπολογιών και να μην λένε ότι ε, το κάνουμε γρήγορα και πρόχειρα. Έχουμε 24 ομάδες εργασίας, διαβάσαμε την αξιολόγηση, μιλήσαμε με 900 ενδιαφερόμενους. Δεν πέσαν αυτά από τον ουρανό και ξαφνικά διαπιστώσαμε μία μέρα ότι πρέπει να γράψουμε ένα πρόγραμμα έρευνας. Όχι, έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, απόψεις και προτάσεις για την διαφορομόρφωση του πρόγραμματος. Μη λέτε λοιπόν το κάναμε γρήγορα και πρόχειρα. Το επαναλαμβάνω. Σε συγκεκριμένους ε, τομείς, τεχνητή νοημοσύνη, κβαντομηχανική κτλ. Έχουμε, θα έλεγα, ένα περιθώριο 2-3 ετών και μπορούμε να διαμορφώσουμε ε, κάποιους τομείς στους οποίους είχαμε ένα πλεονέκτημα. Σε κανέναν από τους τομείς στους οποίους είχαμε πριν από 20 χρόνια ένα προβάδισμα δεν έχουμε πλέον κάποιο περιθώριο. Αν μιλάμε για ε, για υπολογιστέ. υπολογιστές. Αν χρειάζεται δύο χρόνια για να φτιάξουμε μια κοινοπραξία στην ε, Κίνα το χρηματοδοτούν ήδη με 5 δισεκατομμύρια. Οι Αμερικανοί μέσω του στρατού τους επίσης πάνε σε ανάλογη κατεύθυνση. Μη λέμε λοιπόν ότι τα κάνουμε γρήγορα και πρόχειρα. Αν κινηθούμε αργά θα χάσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι να αποφασίσουμε γρήγορα ότι το... και το Κοινοβούλιο να κάνει μια λογική πρόταση και το Συμβούλιο την τελευταία φορά αποφάσισε γρήγορα και καθυστερούσαμε μήνες γιατί δεν μπορούσε να συμφωνήσει το Συμβούλιο κάποια στιγμή. Περιμέναμε μήνες ολόκληρος. Δηλαδή αυτό δεν ήταν ποιότητα, ήταν απλά αργοπορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους δύο εισηγητές ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές. για την πολύ σκληρή δουλειά που έκαναν. Τελειώσαμε το σημείο 5 και 4 και 5. Σημείο 6. Θέσπιση του προγράμματος Invest EU. Ο συγητής είναι ο Σον Κέλλη. Μόλις ήρθε. Ωραία, ευχαριστώ. Και να τονίσω ακόμη μια φορά ότι για το θέμα αυτό και ο εισηγητής παρουσίασε το σχέδιο έκθεσης πριν από τις διακοπές, το οποίο ακριβώς δείχνει ότι η Επιτροπή μας θέλει να επιτυχεί ε, συμφωνία σε αυτήν τη θητεία. Και να πω ότι περνάμε στη συζήτηση. Να λόγω και ο Σόν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Είμαστε... Είμαι συγητής για αυτό το φάκελο. Και φυσικά αυτό έρχεται κατόπιν της επιτυχίας του ΕΦΣΥ και ελπίζουμε το Invest EU να φέρει 50 δισεκατομμύρια προς επενδύσεις ε, στην ε, οικονομία. Έχουμε μεγάλη όθηση στην ανταγωνιστικότητα και στην ευμερία και πιστεύω ότι θα βοηθήσει τις μικρές και μισές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να πετύχουμε τους ε, στόχους για το κλίμα και για την ενέργεια. Και αναφέρομαι και σε αυτά που είπε ο συνάδελφος για το τελευταίο φάκελο και αυτά είναι ιδιαίτερα σχετικά το σχέδιο Γιούλκερ εισήχθη το 2014. Πολλοί είχαν αμφιβολίες, όμως από τότε σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν το Ταμείο InvestEU τώρα θέλει να είναι πιο στοχευμένο στις επενδυτικέ πολιτικές μας και να φέρει μεγέθυνση στις επιχειρήσεις μας και στους τομείς όπου χρειάζεται περισσότερο και χρειάζεται ακόμη παρά την επιτυχία του ΕΦΣΙ. Τα επίπεδα επενδύσεων στην Ένωση είναι κάτω από τα επίπεδα του 2009 ακόμη και ε, σημαντικές, ε, σημαντικά προβλήματα είχαμε για τις οικονομίες μας, τα ανέφερε και ο Κρίστιαν και φυσικά έχουμε και το πρόβλημα του Brexit τώρα το οποίο φέρνει διάφορα σοκ σε πολλά κράτη-μέλη, ακόμη και στις καλύτερες περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με ένα φιλόδοξο μέσο μόχλευσης του κινδύνου για να ενθερύνουμε τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είπατε Πρόεδρε, στη γνωμοδότησή μου έχω επικεντρωθεί σε κάποιες τροποποίησεις της πρότασης Κομισιόν που πιστεύω θα βοηθήσουν για να λειτουργήσει καλύτερα και ότι θα πετύχουμε το στόχο των επενδύσεων. Καταρχήν, κοιτάζω το θέμα της διακυβέρνησης. Θέλω να διασφαλίσω στη διακυβέρνηση ότι υπάρχει δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στην εξέταση των project που θα στηριχτούν μέσω της εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσω ότι υπάρχει κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την, να εφεύρουμε τον τροχό και γι' αυτό προτείνω να ε, προσφύγουμε σε, ε, σε κυβερνητική δομή, κάτι που υπάρχει ήδη για το ΕΦΣΙ. Στην πρόταση της Κομισιόν, τελικά η Κομισιόν μέσω της ε, ομάδα. για τα project θα αποφασίσει αν γίνονται σεβαστέ οι πολιτικέ τη Ένωση. Εγώ όμω έχω εισαγάγει και μια διευθυντική επιτροπή όπου θα υπάρχει εκπροσώπηση από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, άλλου εταίρου ε, και έναν εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η επιτροπή θα διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται το Ταμείο σύμφωνα με τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θέλει να πετύχει την επιτεύξη στρατηγικών στόχων θα υπάρχει και ένα συμβουλευτικό σώμα, έτσι όπως προτείνεται από την Κομισιόν, ε, και θα ε, συμμετέχουν εκεί η Κομισιόν, ε, τα κράτη-μέλη και οι εταίροι εφαρμογής. Θέλουμε να είμαστε πιο διαφανείς ως προς το την απόρριψη project που δεν συνάδουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως μου τόνισαν ότι ε, το scoreboard που προτείνει η Κομισιόν ε, θα πρέπει να εισαχθεί εκ νέου. Το καλωσορίζω αυτό και θα ήθελα να συζητήσω εκ νέου την επανασυγωγή με τους σκιώδεις ως ένα πρόσθετο καθήκον της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής. Έχω επίσης συμπεριλάβει εμπειρογνώμονα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό εδώ να έχουμε την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για να πετύχουμε μέχρι το 2030 τους στόχους για την ενέργεια και το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή έχει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για τη χρήση της ευρωπαϊκής εγγύησης για την επίτευξη των στόχων. Σε ό,τι αφορά την κατανομή τη Ευρωπαϊκή εγγύησης, θέλω να διασφαλίσω έναν ε, σαφή ρόλο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καλωσορίζω την πρόταση να υπάρχει ένας ρόλος για τις εθνικές ε, ε, τράπεζες τι αναπτυξιακέ θα πρέπει να συσταθούν αναπτυξιακές τράπεζες σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα διασφαλίσει καλύτερη γεωγραφική κατανομή στην χρήση των κονδυλίων και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο προσθετικότητα, είναι προσθετικότητα. Είχε εισαχθεί η προσθετικότητα από την Κομισιόν, Όμω δεν υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια δικαίου. Έτσι λοιπόν έχω εισαγαγεί ένα νέο άρθρο για να ορίσουμε τι λέμε, τι εννοούμε με τον όρο προσθετικότητα. Θέλουμε να αντιμετωπιστούν οι αποτυχίες της αγοράς ε, σε κάποιες ε, καταστάσεις επενδύσεων που δεν είναι οι βέλτιστες. Ε, θα πρέπει ε, ουσιαστικά να, δούμε και μια πολύ σημαντική αλλαγή θα είναι, δεν θα ζητά, παραδείγματο χάρη, το ΕΦΣΥ να επενδύσει σε project υψηλού κινδύνου. Οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σήμερα από ό,τι πριν τέσσερα χρόνια. Κάτι ακόμη που θέλω να αναφέρω και ξέρω ότι μακρηγορώ είναι η σημασία ε, του κόμβου συμβουλών. Έχω τροποποιήσει το κείμενο έτσι ώστε ο κόμβο συμβουλών να έχει παρουσία σε κάθε κράτο μέλο. Θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να ενημερώνονται οι πολίτε και επιχειρήσει για τις διαθέσιμες ευκαιρίες ε, προκειμένου να καθοδηγεί τους ετούντες ε, στις διαδικασίες και να υπάρχει ενημέρωση για τα project σε πρώιμο στάδιο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα InvestEU επικεντρώνεται στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει επιχειρήσεις, το 20% της χρηματοδότησης ε, θα πηγαίνει στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, σήμερα, όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον. Το InvestEU ε, απλουστεύει την διαδικασία χρηματοδότησης, γιατί συγχωνεύει κάποια εργαλεία. Επίσης, συμπληρώνει τη χρηματοδότηση, όπως είναι το Innofin και το COSME. Τέλος να πω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συνάδει με τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας ε, για να έχουμε καθαρά ε, κλιματικά και ενεργειακά project και ενεργειακή αποδοτικότητα και στο πλαίσιο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είχα και διάφορες δημόσιες συνεδριάσεις στην εκλογική μου περιφέρεια τα τελευταία δύο χρόνια και κάλεσα τους επιχειρηματίες ε, και τους πολίτες να έρθουν και να θέσουν ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και στην Κομισιόν ε, και πολλοί συμμετείχαν. Όμως είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα για ένα πρόγραμμα που μοχλεύει τον κίνδυνο στα πλαίσια του Invest in You. Ε, με τους κατάλληλους κανόνες μπορούμε να το κάνουμε να πετύχει. Σας ευχαριστώ. Σας ευτυχώς δεν είχαμε μετρήσει το χρόνο ε, και έτσι δεν ξέρουμε πόση ώρα μιλήσατε. Ευχαριστούμε πάντως και όλοι οι τώρα παρακαλώ ο κ. Κόλλοντ. Να ευχαριστώ τον συγγητή, τον Τζον Κέλλη, για την πολύ καλή δουλειά του κατά την προπαρασκευή τη έκθεση και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του τι επόμενε εβδομάδε. Ο κ. Κέλλη ενισχύει την υπάρχουσα νομοθεσία με την έκθεσή του. Υπάρχουν μια σειρά αποθετικά στοιχεία σε αυτά που προτείνει. Με το Invest EU έχουμε τη δυνατότητα αυτό πρέπει να δούμε τι πρέπει να υποστηρίξει πιο στοχοθετημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και με βάση αυτό να καθοδηγήσουμε τι μελλοντικέ επενδύσει. Με τον ε, προκάτω, προκάτω χώρο, με το προηγούμενο πρόγραμμα, δυσκολευτήκαμε να ε, οδηγήσουμε τις επενδύσεις στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ελπίζω, ελπίζω με το InvestEU να φτάσουμε σε μια συμβαστική λύση έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες στις οποίες θα αναφερθώ ε, στις τομείς όπου έχουμε αρμοδιότητα βέβαια και κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι στην καρδιά αυτής της νομοθεσίας. Ε, να ενισχύσουμε τους τρόπους διασύνδεσης της Ευρώπης περαιτέρω, είτε ψηφιακά είτε μέσω μοντέρνων υποδομών. Το είπε και ο Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασύνδεση στην Ευρώπη. Η έρευνα στους, ε, στις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες για να επελευθούν οι μεγαλύτερες προκλήσεις προς την, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, στην αγορά και αντιμετώπιση τη περιβαλλοντική αλλαγή ε, μέσω νέων τεχνολογιών και νέων επενδύσεων για να μπορέσουμε να, να προωθήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τους Ευρωπαίους. Αν, αναμένω με ανυπομονησία τη συνεργασία μας κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Από τους πράσινους τώρα, η κυρία Μέτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Κέλλη, ε, για το έργο του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επενδύσεις αυτή τη στιγμή σε μια στιγμή, σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περικοπών. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις για να μπορέσουμε να αργαστήσουμε ε, τις υποδομές, να καταρτήσουμε τους εργαζομένους, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και βεβαίως ε, να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Η InvestEU πρέπει να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει δυνατότητα στους εργαζόμενους, στους πολίτες ε, να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη κατάρτιση και επανακατάρτιση για να μπορούν να συμμετάσχουν στην οικολογική μετάβαση. Θα πρέπει να φτάσουμε επίσης σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα το 2050 το αργότερο και πρέπει το InvestEU να είναι ένα ε, εργαλείο για να φτάσουμε σε αυτήν τη μετάβαση. Δεν θα εκπλαγείτε βέβαια αν επιμείνω ε, στις τροπολογίες μου για υψηλότερους στόχους ό,τι αφορά τις δαπάνες ε, για το περιβάλλον στο InvestEU. Θέλουμε να υπάρξει μια οριζόντια προσέγγιση στο, σύστημα ζήτημα του περιβάλλοντος σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις μας στα πλαίσια των, της Συμφωνίας των Παρισίων. Μία από τις τέσσερις πολιτικές του InvestEU για το μιλάμε για κοινωνική, ε, περιβαλλοντική, κλιματική ε, βιωσιμότητα, αλλά δεν γίνεται μόνο με ένα τέταρτο των χρημάτων να πετύχουμε ε, τους στόχους μας, ενώ μετά τα τρία τέταρτα των χρημάτων να επιτείνουμε τα, τα φαινόμενα μόλυνσης. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλε τι πλευρέ εδώ. Χαίρομαι για την ορισμό σα, για την προσθετικότητα. Για την Θέλουμε να προωθήσουμε εδώ project τα οποία δεν θα, δεν θα τύχαν χρηματοδότηση αλλιώ. Πρέπει να φτάσουν τα χρήματα στον αποδέκτη του, πρέπει να, να χρησιμεύσουν για τον σκοπό για τον οποίο το διαθέτουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον ορισμό αυτό και να υπογραμμίσουμε τη μακρο, το μακροπρόθεσμα κοινωνικά ωφέλη από τον project αυτόν. Υπάρχει και μια άλλη προτεραιότητα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε διαφανείς και ε, κυβερνητικές δομές που να λογοδοτούν ε, στις ε, επιτροπές επενδύσεων, στις, στις, ε, στα διευθυντικά συμβούλια και πρέπει να είναι ισορροπημένα σε αυτέ οι αρχέ και σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων και πρέπει να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια που θα καθορίζεται, όπως είπε ο κ. Σκέλη, σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Επίσης χαίρομαι για τις τροπολογίες ό,τι αφορά την περιφερειακή ισορροπία, έτσι ώστε τα, τα χρήματα αυτά να είναι διαθέσιμα για όλες τις περιφέρειες, όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος ε, του Advisory Hub, έτσι ώστε τα μικρότερα project να μπορούν να συμπτύσσονται, να δημιουργούν μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια και να είναι έτσι ε, πιο εύκολο να χρηματοδοτηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εγώ αναμένω με ανυπομονησία τη συνεργασία μου μαζί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την Γκουή, κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον εισηγητή τον κύριο Κέλλη για το για το σχέδιο νομοδότησης, γιατί αφορά πραγματικά σε έναν πολύ σημαντικό φάκελο, στον οποίο θέλω και εγώ να συμβάλλω ε, επικοδομητικά. Αλλά βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ επιτυχία ούτε καλωσορίζω την μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τη δημιουργία του νέου προγράμματος Investium Οι πληροφορίες ε, σχετικά με τις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και την πορεία υλοποίηση των έργων του μέχρι σήμερα δεν τεκπηριώνουν αν και κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους του και αν δικαιολογείται ένα ειδικό καθεστώς στήριξης των επενδύσεων. Ακόμη και αν δεχθούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Δεκάτου 17 το πραγματικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του και σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια τη ιδιαίτερα βιαστική διαδικασία για τη χρονική και οικονομική τη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων το Φεβρουάριο του 2017. Συμφωνώ στην των υποψήφιων έργων. Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του ορισμού τη στο παρόν νομοθέτημα και δεν επαρκεί η παραπομπή του δημοσιονομικού κανονισμού. Απαιτείται σοβαρό εξορθολογισμό τη δομή διακυβέρνηση του Ιβέστιου ενίσχυση της διαφάνειας το μοντέλο της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των στρατηγικών αποφάσεων, ενώ αποκλεί την απαραίτητη κατά την άποψή μου εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κλείνοντα, είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυση τη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγηση των έργων και επιλογή έχουν προσωπικό χαρακτήρα και να υλοποιηθούν μέσω των λοιπόν χρηματοδοτικών Δεν θεωρώ απαραίτητη την οργάνων στη διαδικασία επιλογής καθότι θα επιφέρει καθυστέρηση και θα εντείνει στην πολυπλοκότητα του όλου, ε, του όλου διαβήματος. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να, να και να κλείσω θα προτείνω όσον αφορά στην επιπλήρωση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την Thank you very much, madam. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ευθυντή κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ. Όπως και το ΕΦΣΗ παρουσίασε διάφορα σημεία επίκρισης ε, και εδώ ισχύει το ίδιο. Σίγουρα ο στόχος ενός νέου προγράμματος επένδυσης